Κύριε Επίτροπε, έχετε την δυνατότητα να μιλήσετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θεωρώ ότι τελευταίες ε, θα μπορούσαν να είναι μια ένδειξη για των καταληκτικών μου λόγων. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ένα πολύ θετικό βίωμα ε, και πρώτη φορά είχα την αίσθηση ότι είναι λιγότερο μια κρόαση και περισσότερο μια ανταλλαγή απόψεων. Και αυτός ακριβώς είναι και ο τρόπος που βλέπω εγώ τα πράγματα και που θέλω να τα αντιμετωπίσω μελλοντικά. Να έχουμε έναν κοινό, να έχουμε έναν διάλογο, ούτε ώστε να καταλήξουμε σε μια θετική έκβαση. Βεβαίω δεν είναι δυνατό να συμφωνούμε 100% σε όλα. Ε, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό στο πλαίσιο μιας πραγματικής δημοκρατίας, αλλά δεν είναι ούτε τραγικό. Σημαντικό είναι να μας διαπικινεί βούληση να πετύχουμε κάτι προς όφελος των πολιτών μας. Εγώ θα φροντίσω το ώστε το ευρωπαϊκό εγχείρημα να προχωρήσει και ε, να θα προσπαθήσω να κατοχυρώσω τα ευρωπαϊκά μας ε, συμφέροντα και ε, να δώσω τη δική μου συμβολή στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας ούτως ώστε η ζωή να γίνει πιο ασφαλής, να έχει περισσότερες ε, προοπτικές ε, στο μέλλον, να υπάρξει για τις χώρες αυτές ε, της γειτονία, να έχουν μια προοπτική τόσο ίδιος και τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους. Ε, ελπίζω να υπάρξει τόσο στο στερκό της Ευρώπης όσο και στις γειτονικέ χώρες μια ε, τεράστια δυνατότητα διακίνησης, μετακίνησης των πολιτών ε, και να νομίζω ότι αν μπορέσουμε τα επόμενα πέντε χρόνια να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι μεγάλη η δική μας συμβολή και είμαι διατεθειμένος να δεσμευτώ προσιλωμένο σε αυτό το στόχο και βεβαίως αναμένω και τη δική σας υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Βλέπετε ότι η Επιτροπή αυτή είναι μια φιλικά διακείμενη Επιτροπή, αλλιώς δεν θα μπορούσατε να απολαύσετε αυτό το θερμό χειροκρότημα, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να γίνουμε και λιγότερο φιλικοί συν το χρόνο. Εγώ προσωπικά αξιολογώ το χειροκρότημα των συναδέλφων σαν μια θετική ένδειξη της αξιολόγησης ε, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις που δώσατε. Βεβαίως δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις που δόθηκαν και δεν θα ήταν καλό να ήταν όλοι ικανοποιημένοι, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για μια μελλοντική συνεργασία και στην περίπτωση που συντάξουμε πράγματι μια ε, φιλική επιστολή ε, θα ήθελα να μας ευχηθώ καλή συνεργασία οι συντονιστές θα συναντηθούν ε, για να συντάξουν αυτή την φιλική επιστολή.